ζήτησε θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. Έκθεση της κυρίας Αλφάνο για το οργανωμένο έγκλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτρια για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την από τη συνεργασία με τους κυρίους, τους κυρίους Γιακολίνο, Κροτσέτα, Μπέρτ, Άλμπρεχτ και Ντε Ιόγκ. Είναι τέσσερι ισχυώδεις συζητητές από τι άλλε πολιτικές ομάδες. Το οργανωμένο έγκλημα και οι μαφίες αποτελούν μια βασική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε ένα επίσημο κείμενο στις μαφίες ε, και στις ε, διεθνικούς, διεθνικούς τρόπους αντιμετώπισης τους. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο οργανωμένο έγκλημα και στις μαφίες, διότι όπως λέει η Ευρωπολ έχουμε οργανωμένες εγκληματικές μεταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πλήττουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους θεσμούς. Χρειάζονται συντονισμένες μέθοδοι παρέμβαση. Μία θεραπεία η οποία θα πρέπει να έχει να κάνει με, την, με τον ακού, με αυτούς που αντιμετωπίζουν κάθε μέρα το οργανωμένο έγκλημα, ε, ε, νομικούς εγκληματολόγους, νομικούς οι οποίοι εργάστηκαν για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα ζητήματα και που με αυτοθυσία εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη στον αγώνα τους κατά των εγκληματικών οργανώσεων. Το κέρδος είναι το κίνητρο των εγκληματικών οργανώσεων. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως πρώτη προτεραιότητα λέμε ότι θα πρέπει να κατάσχουμε όλες τις περιουσίες που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα. Πρέπει να δούμε με ιδιαίτερα ενδιαφέρον την πρόταση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά είναι ένα κόρπους γιούρις για την κατάσχεση των εγκληματικών περιουσιών ή μάλλον των περιουσιών που γεννήθηκαν από το έγκλημα. Θέλουμε εμείς ευρωπαϊκούς κανόνες για διευρυμένη κατάσχεση ακόμη και όταν δεν έχουμε καταδίκη θα πρέπει να κατάσχονται και οι διοκτησίες οι οποίες ανήκουν σε ε, άτομα ε, μαϊμούδες που δανείζουν το όνομά τους στους εγκληματίες. Αυτό θα ήταν μια καλή προσπάθεια. Εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω ποιες απαιτήσει έχουμε. Εναρμόνιση των διατάξεων για το οργανωμένο έγκλημα, μεγαλύτερη προστασία των θύματων, ενιαία διαπίστωση των, μαφιών, στις, ε, στα κράτη-μέλη, συνεργασία της Eurojust, της Europol, της Olaf με τα εθνικά κράτη, αμοιβαία αναγνώριση των, νομικών, των δικαστικών αποφάσεων, διαφάνεια και πρόληψη για να αποφύγουμε οι δημόσιες, ε, τα δημόσια κονδύλια να πέφτουν στα χέρια των εγκληματιών. Να αποφύγουμε την ανακύκλωση του βρωμικού χρήματος θα πρέπει να μην επιτρέπουμε σε υπόπτους ε, ή καταδικασμένους να είναι υποψήφοι σε εκλογές. Εμείς ε, θέλουμε να μην είναι μόνο λόγια, κύριε Επίτροπε, αυτά που θα εγκρίνουμε. Εμείς θα θέλαμε να περάσουμε στα έργα, ευθυγραμμιζόμενοι με τις συνθήκε και με τον απόλυτο σεβασμό της Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου Οι βασικοί κριτές της προάσπισης των ελευθεριών των πολιτών είναι τα εθνικά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα θέλαμε να ληφθεί υπόψη η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το τελευταίο που είναι και ίσως το πιο σημαντικό. Εγώ θα ήθελα αυτό το πρώτο βήμα που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα θύματα του οργανωμένου εγκλήματος ε, σε όλους εκείνους ε, οι οποίοι δεν ε, κάμφθησαν ηθικά. Ελπίζω αύριο λοιπόν να δώσουμε ένα θετικό μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Αλφάνο. Ο κύριος Γιακολίνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την ε, εισηγήτρια την κυρία Αλφάνο η οποία δίνει μια σημαντική όθηση σε ένα σημαντικό μέτρο η οποία συνεισφέρει σημαντικά σε... και μας δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο για να αντιμετωπίζουμε καλύτερα και πιο αποφασιστικά όλα τα φαινόμενα μαθίας και οργανωμένου εγκλήματος με αυτό το μέτρο αλλά κυρίως με τις προτάσεις που θα προωθήσει η Κομισιόν δεν θα έχουμε τα, τους τωρινούς φραγμούς για να μπορέσουμε να κατασχέσουμε τις περιουσίες των μαπιόζων και να μπορέσουμε να, τους, να διαφυλάσσουμε αυστηρή φυλάκιση για όσους έχουν σημαδευτεί με τέτοια εγκλήματα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε τους συνεργάτες με τη δικαιοσύνη, να έχουμε αμοιβαία δικαστική συνεργασία, να έχουμε μία πρωτοποριακή νομοθεσία υπέρ των τιμίων πολιτών, των τιμίων επιχειρηματιών και να μπορέσουμε να ανταμείψουμε πια και ηθικά αυτούς που δεν έσκυψαν το κεφάλι τους στη μαφία αλλά περήφανα τις αντιστάθηκαν. Ευχαριστώ η κυρία Ζαμπόρσκα. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πίτροπε, η προστασία όλων των πολιτών της ευρωπαϊκή Ένωσης από δραστηριότητες οργανωμένου εγκλήματος έχει τεράστια σημασία. Όμως το πιο σημαντικό είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τα παιδιά και οι νέοι, οι νεαροί και οι νέοι άνθρωποι. Η προστασία ακριβώς παιδιών δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συνεργασία με τους γονείς τους. Πριν από χρόνια ανέλαβα την πρωτοβουλία μιας ευρωπαϊκής εκστρατείας με ερώτημα. Ξέρετε που είναι τα παιδιά σας, που βρίσκεται το παιδί σας ή βρίσκονται τα παιδιά σας τώρα. Και με ένα φυλάδιο ενημερωνόντουσαν οι πολίτες, οι γονείς, ποιες ήταν οι κυριότερες απειλές στο, εις βάρος των παιδιών τους. Συνάντησα τρεις επιτρόπους από τότε μέχρι σήμερα. Τόσα χρόνια πέρασαν και εξακολουθούν να υφίστανται απειλές για τα παιδιά. παρόλα αυτά δεν βρήκα καμιά θετική ανταπόκριση από πλευράς επιτρόπων για αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ η κυρία Κώστα. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια Αλφάνο για τη σημαντική της έκθεση που αποτελεί ένα βασικό σημείο αναφοράς για τη δράση του Κοινοβουλίου γύρω από ένα θέμα το οποίο αποτελεί σήμερα νέα και ενισχυμένη αρμοδιότητα με την συνθήκη της Λισαβόνας αλλά και το θέμα της αντιμετώπισης ε, των ε, μαφιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση με Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με ενιοποίηση νομοθεσιών στα κράτη-μέλη. Όλα αυτά είναι θεμελιώδη. Εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι ορισμένες από τις προτάσεις μου ελήφθησαν υπόψη για, τον, για την πρόθεση ε, του ρόλου των ενώσεων των οικογενειών των θυμάτων. Επίσης μια ολιστική αντιμετώπιση για το θέμα της διακίνησης ανηλίκων. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω ακόμη περισσότερο ότι οι γυναίκες και οι ανήλικοι είναι το μεγαλύτερο μέρος των θυμάτων των εγκληματικών οργανώσεων. Πρέπει να υπάρχει μια ειδική στράτευση, μια υποστήριξη και προστασία των γυναικών που είναι θύματα όλης αυτής της βίας. Ακόμη και γυναίκες οι οποίες βρίσκονται μέσα σε αυτές τις μαφιόζικες οικογένειες και αντιστέκονται στην ανηθικότητα. Επίσης θέλω να τονίσω τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην εισαγγελία στην, ε, ε, στο, στο δικαστικό σώμα αλλά και στα σχολεία οι καθηγήτριες οι οποίες προσπαθούν να αλλάξουν την οτροπία των παιδιών. Πλατσίκοβα, σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η καταπολέψη του οργανωμένου εγκλήματος ε, είναι μέρος και τμήμα τη δικαστική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και μία από τι προτεραιότητε όσον αφορά το συντονισμό που πρέπει να επιτευχθεί και να βελτιωθεί από τα κράτη-μέλη. Η νομοθεσία, το νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να βελτιωθεί σε εκείνου του τομεί και τα μέσα που είναι τα πιο αποτελεσματικά και οι πιο αποτελεσματικοί για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο και των μαφιόζων. Υποστηρίζω την ιδέα τη κυρία Σόνια Αλφάνο να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία να υποστηριχθεί η δίμευση, η των ε, περιουσιακών στοιχείων και ε, χρημάτων και κερδών από τέτοιες ε, εγκληματικές δραστηριότητες. Ε, επίσης είμαι υπέρ της ιδέας του να αναδιανέμονται τα, χρήματα τα οποία θα έχουν κατασχεθεί ή δημευθεί και να μπορούν έτσι να χρησιμοποιηθούν πιο αποτελεσματικά και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα για την προστασία μαρτύρων σε ένα πλαίσιο προστασίας μαρτύρων. Ευχαριστώ. Άλμπρεχτ παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρία Ρέντινγκ, Επίτροπε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, συνάδελφοι, σε αυτό το σημείο έχουμε ένα καλό συμβιβασμό που πετύχαμε θα έλεγα. Και πάλι πρώτα ευχαριστώ θερμά την κυρία συνάδελφο Αλφάνο για, αυτό, για αυτή την έκθεση για την καταπολέμηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων. Ω πράσινη υποστηρίζουμε αυτή την έκθεση και είναι σημαντικό να σημειωθεί πρόοδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει και αντίστοιχε προτάσει σε σχέση με αυτό το θέμα και είναι καλό, είναι θετικό ότι ω Ευρωκοινοβούλιο μπορούμε να πούμε τώρα προς τα που πρέπει να πορευτούμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσουμε. Δεν συμφωνούμε με όλες τις προτάσεις, αλλά η περαιτέρω συζήτηση θα καταδείξει τι πρέπει να γίνει. Η έκκλησή μου απευθύνεται πρώτα στο Συμβούλιο και στα κράτη-μέλη, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε το εξή. Μεγαλύτερη συνεργασία θα είναι δυνατή και εφικτή όταν θα έχουμε πρότυπα δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας που θα καταλήγουν σε κοινά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινοτικά πρότυπα. Και υπερβολικά είναι είναι εναντίον πολλές φορές στα κράτη-μέλη της ενιοποίησης ε, του ενιαίου πλαισίου αυτών των δραστηριοτήτων. Όταν όμως θέλουμε να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα έχει τεράστια σημασία να γίνεται αυτό. Ευχαριστώ. Grazie, la parola all'onorevole Pasca. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τον λόγο, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε από πλευράς του εισηγητού του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Ντίκ Μαρτί, όταν δημοσιοποίησε την έκθεσή του πέρσι για τις δολοφονίες στο Κωσυφοπέδιο, ο κύριος Μάρτι του Συμβουλίου της Ευρώπης λέει ότι ο Χασίμ Θάση, πρωθυπουργός του Κωσυφοπεδίου αυτή τη στιγμή, είναι, ήταν, λέει, κατά τη διάρκεια του τέλους της δεκαετίας του 90, αρχηγός μιας συμμορίας που δολοφονούσε και ασχολείται με εμπόριο ανθρωπίνων οργάνων. Ξεκίνησε μια έρευνα για αυτές τις ε, ε, για αυτούς τους ισχυρισμούς της έκθεσης ε, Μάρτιν. Θεωρούμε ότι αυτά τα θέματα είναι τεράστια σημασία, είναι πολύ σοβαρά. Δεν πρέπει μόνο να βασιζόμαστε στην, στην αρρωγή των αρχών του Κωσυφοπεδίου και του, των δικαστικών αρχών ιδιαίτερα όταν έχουμε και πρόσφατες δολοφονίες γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για τα Δυτικά Βαλκάνια Ευχαριστώ Η Επίτροπος Ρέντινγκ έχει το λόγο Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Ευχαριστούμε κυρία Αλφάνο την πληρέστατη την έκθεσή σα. Ο μακρύτατο κατάλογο των συστάσεων σίγουρα θα αποτελέσει πηγή έμπνευση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι μελλοντικέ εργασίε τη. Η οργανωμένη εγκληματικότητα καλύπτει διάφορου τομεί παράνομη και έκνομη δραστηριότητε και είναι παγκόσμιο φαινόμενο όπω και η καταπολέμηση τη οργανωμένη εγκληματικότητα. Άρα δεν ξαφνιαζόμαστε που ε, ασχολείστε με τομείς πέρα από τις εσωτερικές υποθέσεις τη συστάσεις της. Οι προτάσεις θα μας βοηθήσουν ε, ούτως ώστε να εντάξουμε την καταπολέμηση οργανωμένης εγκληματικότητας σε άλλες πολιτικές όπως οι σχέσεις μας με τρίτες χώρες ε, έκκληση προς τα κράτη-μέλη να κυρώσουν τα επιστάμενα νομικά μέσα που είναι η δομική λύθη για το οικοδόμημα. Επίσης ε, θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά ε, διάφορες ε, νομικές πράξεις και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους εταίρους μας σχετικά με τη μεταγραφή της απόφασης πλαίσιο για την καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας θα ε, μελέτη ώστε να έχουμε μια σαφή και σφαιρική εικόνα της κατάστασης. Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οργανωμένη εγκληματικότητα έχει στρατηγικό χαρακτήρα και βασίζεται σε κοινού στόχους. Αυτό αναφέρεται ε, στην ε, ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Νοεμβρίου του 2010 σχετικά με τη, τους εσωτερικούς στρατηγικούς στόχους και μια ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την εσωτερική ασφάλεια που θα έχετε ε, περισσότερες λεπτομέρειες. Ένας από τους βασικούς στόχους είναι η καταπολέμηση της οργανωμένης εγκληματικότητας, να εκριζώσουμε την ε, κινητήριο δύναμη επίσης να, ε, της εγκληματικότητας, επίσης ε, η διαχείριση των ε, χρημάτων προκύπτουν από παράνομες δραστηριότητες. Σχάτως εγκρίναμε και ένα πακέτο κατά της διαφθοράς, χάρη στο οποίο θα αναλυθούν σοβαρότερες δεσμεύσεις και επίπεδο κρατών μελών για να εκριζωθεί αυτό το φαινόμενο. Ε, η κατάσχεση και η ανάκτηση των κερδών ε, παράνομης δραστηριότητας είναι βασική ε, συνιστός αυτής της προσπάθειας και προετοιμάζουμε νέα νομοθετική πρόταση που θα αντικαταστήσει τα εφιστάμενα μέσα και θα ενισχύσει την δυνατότητα των κρατών μελών να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία. Επίσης, ε, η ε, οδηγία περί οικονομικών πληροφοριών θα μας οδηγήσει σε εκπόνηση στρατηγική από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2012. Η Europol και η Eurojust επίση εξακολουθούν να έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί υποστηρίζουν την αστυνομική και τη δικαστική συνεργασία και έχουν σημειώσει πολλές επιτυχίες πρόσφατα ε, με το θέμα της παιδικής πορνογραφίας και το εμπόριο παιδιών, διάφορες επιτυχίες που σημειώθηκαν ε, καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα των οργανισμών και θα πρέπει να εξετάσουμε τρόπους ώστε να ενισχύσουμε και ίσως και να διευρύνουμε τη δράση τους στο μέλλον. Ε, Κυρία Αλφάνο, έχετε συμπεριλάβει και άλλα στοιχεία και άλλες προτάσεις στην έκθεσή σας. Πολύ συγκεκριμένα θα επανεξετάσουμε όλα τα μέτρα που προτείνετε. Αύριο συγκεκριμένα η Επιτροπή θα υποβάλει μία ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή αντίδραση ε, ως προς τα αρκωτικά. Και αυτό θα εγγράφεται στη συνολική στρατηγική Καταπολέμησης ε, ε, του εμπορίου και της κατάχρησης ναρκωτικών. Ελπίζουμε ότι θα συνεχίσετε να μας βοηθάτε όχι μόνο με εκθέσεις αλλά και με συγκεκριμένες δράσεις γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πέρα στη συζήτηση θα ψηφίσουμε αύριο στις 12.30. και Τώρα τελευταίο έκθεση του κύριου Πρέντα.